Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Περιμέναμε λίγο να καθίσετε. Μπορούμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση της Συνόδου της Ολομέλειας και θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος άρθρο 154. Έχουμε την πρώτη.